Η Γεια σα. Καλησπέρα σα, Επαναλαμβάνετε η συνεδρίαση. Έχετε τα πρακτικά τη χθεσινή συνεδρίασης στη διάθεσή σα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσει, Αν όχι, εγκρίνονται τα χθεσινά πρακτικά.